γιατί μου φάνηκε ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ε, δουλειά που έκανε. Αυτό είναι σημαντικό για μένα να το υπογραμμίσω. Ε, να έχει ένας αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τόσο στενές σχέσεις με αυτή το κοινοβούλιο στο οποίο υπήρξα ε, και συνεργάστηκα επί 15 χρόνια. Όσον αφορά την βιομηχανική κατάσταση, την κατάσταση της βιομηχανίας, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα πράγματα. Η συζήτηση αυτή που γίνεται σήμερα το βράδυ είναι πολύ σημαντική για όλους. Ευτυχώς, μετά από χρόνια που η Ευρώπη στόχευσε περισσότερο προς τις υπηρεσίες και ε, τα χρηματοοικονομικά ζητήματα σαν την καρδιά της οικονομίας, ευτυχώς σήμερα η Ευρώπη αρχίζει να συζητάει την σημασία ε, ενός σύγχρονου ανταγωνιστικού βιομηχανικού συστήματος, ενός συστήματος πράσινου, κατάλληλου ε, να πρωταγωνιστήσει στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, ε, στα πλαίσια μιας ανάπτυξης που θα μπορέσει να δημιουργήσει απασχόληση και που θα μπορέσει να μας κάνει να κερδίσουμε τη μεγάλη αυτή πρόκληση απέναντι στην κρίση. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή της, ε, της δεύτερης θητείας του Μπαρόζο άρχισε στα πλαίσια του ορίζοντα Ευρώπη 2020 να υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της βιομηχανικής πολιτικής. Δεν είναι η βιομηχανική πολιτική που είχαμε πριν από 20-30 χρόνια, μια σύγχρονη, μια μοντέρνα βιομηχανική πολιτική. Για να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τα όσα χάσαμε τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, σήμερα τα στοιχεία για την βιομηχανική παραγωγή δείχνουν μια υποχώρηση της τάξης του 2% και 1% ε, χαμηλότερο από την κορυφή που είχαμε φτάσει το 2008. Διαφοροποιείται βέβαια ανακράτο και ανακλάδο η κατάσταση αυτή, αλλά αναμφίβολα όλη η ευρωπαϊκή βιομηχανία πλήττεται. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιου τρόπου να φέρουμε την αλλαγή. Ξέρετε πως έχω, είχα διοργανώσει μια μεγάλη εκδήλωση πριν από ένα περίπου έτος στις Βρυξέλλες που είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη και πώς αυτή μπορεί να συνδεθεί ε, με την ε, βιομηχανική μας πολιτική. Είχαμε καλέσει τον Τζέρμι Ρίφκιντ μάλιστα ε, για να κάνει μια παρουσίαση. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουν τα κράτη-μέλη. Και κάποιοι είναι, έχουν καλύτερες αποδόσεις από άλλους. Η Σλοβακία, για παράδειγμα. 18,7% αύξηση σε αιτήσια βάθηση. Η Λιθουανή. Οι επίσης εξαιρετικές επιδόσεις. Αλλά έχουμε την Κύπρο, για παράδειγμα, την Ιταλία, την Ισπανία, που αντιμετωπίζουν πολύ δυσκολότερες καταστάσεις η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη, η Γερμανία, που είχε μία ε, ανάκαμψη, σήμερα αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες. Για τον κλάδο πρέπει να σας πω πως ε, ε, στις κλωστιφεροντουργίες, στα έπιπλα, στην αυτοβιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, στην βιομηχανία πλαστικών, στη χημική βιομηχανία, στα ναυπηγεία. Το 2012 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. παντού είχαμε προβλήματα. Έχουμε και ομάδες εργασίας υψηλού επίπεδου για την αυτοκινητοβιομηχανία, για τη χαλιβουργία, για τις κατασκευαστικές, για τα ναυπηγεία και εκεί διαπιστώνουμε προβλήματα. Ξεκίνησε η κάμψη στην ανεργία, στην απασχόληση το 2012, μετά το 2011. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση, πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις χάθηκαν ε, στη βιομηχανία. Τεράστιο ποσοστό, γύρω στο 10%. Το 2010, τελευταίο τρίμηνο, έχει αυξηθεί η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω αναδιαρθρώσεων. 2.674 αναδιαρθρώσεις που οδήγησαν σε απώλεια 74.560 ε, θέσεων εργασίας και αυτό κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία και ε, στις κατασκευαστικές. Η ανάκαμψη στην Ευρώπη είναι ανίσχυρη ε, και πρέπει να σας πω πως δεν ήταν η αναμενόμενη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δράσουμε αμέσως. Η παγκοσμιοποίηση σημαίνει πως έχουμε μετεγκαταστάσει σε άλλα κομμάτια του κόσμου. Η Κίνα αύξησε 7,7% τη δική της συμβολή στην παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή. Ξεπερνά λοιπόν ε, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το παγκόσμιο εμπόριο από το 17,3% πέσαμε στο 16% του μεριδίου παγκοσμίου εμπορίου. Αυτό το παρουσιάσαμε και τον Οκτώβριο με την ενημερωμένη βιομηχανική πολιτική που θέτει ένα σαφή στόχο. Μία νέα εκ νέου ε, βιομηχανοποίηση της Ευρώπης με 20% ανάπτυξη του ΑΕΠ σε σχέση με το 15% συμμετοχής βιομηχανίας σήμερα. Δεν μιλάμε μόνο για αριθμητικά στοιχεία. Θα πρέπει να έχουμε και τις αντίστοιχες πολιτικές που θα μας επιτρέψουν να καταφέρουμε αυτούς τους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε να ε, εστιάσει την προσοχή της σε έξι βασικές αγορές που μπορεί να επηρεάσουν και τις αναδυόμενες βιομηχανικές αγορές και τις παραδοσιακές βιομηχανικές αγορές της Ευρώπης. Αυτές οι έξι αγορές είναι τεχνολογία, αηφόρος ε, κατασκευή, ε, κατασκευαστικό κλάδος, βιοοικονομία, καθαρά οχήματα και ευφυής χρήση ενέργειας. Στην Γκρενόμπλα της Γαλλίας μεθαύριο θα γίνει και μία σύνοδος πολύ σημαντική με τους υπουργούς βιομηχανίας ε, που θα συνεδριάσουν με ένα κέντρο αριστείας, το ερευνητικό κέντρο της, Ευρω... της Η Task Force που προ ετοιμάζει τον οδικό χάρτη ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη βιομηχανική πολιτική. Σύντομα θα δημοσιεύσει τα πορίσματά της έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών ε, και βιομηχανίας. Έχουμε λοιπόν οριζόντιους στόχους και παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στη βιομηχανία, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε στοχευμένα προγράμματα δράσης. Μίλησα για την αυτοκίνητο βιομηχανία για την οποία έχουμε εγκρίνει στις 8 Νοεμβρίου του 12 ένα σχέδιο δράσης εν ώψη του 2020 για να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του κλάδου που προτείνουμε διάφορες δράσεις στοχευμένους, στοχευμένες για να διαχειριστούμε τις διορθωτικές αλλαγές που σημειώνονται στον κλάδο. Αυτό ισχύει και για τη χαλιβουργία. Ε, ένας ε, γύρω στο τραπέζι σε υψηλό επίπεδο θα συνεδριάσει για τρίτη φορά ε, στις 12 Φεβρουαρίου. Θα τα διαβάσατε άλλωστε στον τύπο. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ε, αυτή την συνάντηση. Η Αρσελόν Μιτάλ, για παράδειγμα, ε, θα έρθει και αρκετοί υπουργοί βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουν τα θέματα του Χάλιβα και θα πρέπει να ξεκινήσουμε και χαίρομαι που το κάνει και με στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβόλιο θα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε ποια είναι η ανάγκη του να έχουμε και ένα συμβούλιο ανταγωνιστικότητας όπου θα μπορούσαμε να συζητάμε βιομηχανική πολιτική και συγγενή θέματα. Δηλαδή, Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Βιομηχανίας, Παύλα Βιομηχανίας. Έκανα ένα πείραμα σχετικά στις 9 Δεκεμβρίου Προσκάλεσε σε γεύμα εργασία στι Βρυξέλλε όλου του υπουργού βιομηχανία για να συζητήσουμε μαζί άτυπα. Αλλά μόνο του υπουργού, Όχι του πρέσβεις. Για να συζητήσουμε θέματα βιομηχανίας, ε, βιομηχανικής φύσης, για παράδειγμα κρίση ε, στην αυτοκινητοβιομηχανία και αν μπορούμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε εκεί τις προκλήσεις. Και μετά στις 10 Δεκεμβρίου έγινε και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και το Συμβούλιο πήγε πολύ καλά. Ακριβώς γιατί είχε γίνει αυτή η πραγματική συνεδρίαση, το πραγματικό Συμβούλιο των Υπουργών Βιομηχανίας την προηγούμενη. Γιατί δυστυχώ το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα πολλέ φορέ μετατρέπεται σε κορεπέρ, όπου έχουμε ε, μόνο πρέσβει ε, και δεν έχουμε υπουργού εκεί είναι δύσκολο να πάρεις αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο, εάν δεν υπάρχουν οι πολιτικοί υπεύθυνοι των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ για μία φορά ακόμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας στηρίζει και που μας σπρώχνει να αποκτήσουμε ένα πραγματικό συμβόλιο βιομηχανίας με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις έτσι ώστε να έχουμε μια νέα σύγχρονη ανταγωνιστική βιομηχανική πολιτική και ευχαριστώ και το Κοινοβούλιο για τη δέσμευση που δείχνει σήμερα, για τη συζήτηση που γίνεται, που είναι σημαντικότατη, πολύ ενδιαφέρουσα για μένα. Εγώ δεν πιστεύω πως θα γίνει η νέα βιομηχανική επανάσταση χωρίς την πραγματική συμβολή του Κοινοβουλίου σας και των συμπολιτών μας. Θα πρέπει μαζί να αξιολογήσουμε μια στρατηγική για την ε, επαναβιομηχανοποίηση με πράσινο τρόπο της Ευρώπης, με σύγχρονο τρόπο, για να κερδίσουν οι εταιρείε αυτή την πρόκληση. Και αυτό δεν αποτελεί όνειρο, είναι στόχος, τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε. Για μια φορά ακόμα σας ευχαριστώ ε, για τη δέσμευση που έχετε δείξει και με την οποία στηρίζετε αυτή τη νέα βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Κρόστη αυτό ΕΛΚ πρώτη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι ένα τεράστιο έργο που έχουμε μπροστά μας σε αυτή τη διαδικασία ε, νέου εκβιομηχάνησης της Ευρώπης η χαλιβουργία έφυγε ήδη στην Ινδία, ε, άλλες βιομηχανίες στην Κορέα, η αυτοκινητομηχανία διαχέθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, η φάρμακοβιομηχανία προς τις ΗΠΑ για να ξεφύγει από την πολύ αυστηρή ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία, η πυρηνική βιομηχανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κίνα και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυτή η βιομηχανική κρίση που φύγει ε, πολύ τεχνολογικούς τομείς. Ε, αυτό έχει πολλές αιτίες. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη χαλιβουργία που παραμένει ένας ε, τομέα κλειδί για την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ε, είναι θύμα των αδυναμιών τη. Δεν είναι αρκετά παγκοσμιοποιημένη. Υφίσταται τι επιπτώσει των διακοιμάσεων των τιμών, του ισχυρού ανταγωνισμού αυξάνεται η Κίνα που γίνεται ε, ο, ο, πρωταγωνιστής του τομέα αυτού ε, παγκοσμίω και διάφορες ε, άλλες αναδυόμενες χώρες. Ε, οι, βιομηχανικές οι οικογενικές επιχειρήσεις έδωσαν τη θέση τους σε μεγάλες πολυεθνικές. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξουμε παγκόσμια πρότυπα. Πρέπει να προβλέψουμε στρατηγικές επενδύσεις και να αποκτήσουμε την ικανότητα να τις χρηματοδοτήσουμε και χάρη και στη δημόσια υποστήριξη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, η Κορέα το κάνουν. Γιατί όχι και εμείς. Αυτό απαιτεί να ε, προσαρμοστούν οι κανόνες μας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, ούτως ώστε να συνεχίσουμε να παίζουμε το ρόλο του εγγυητή ε, μεταξύ των κρατών μελών, υποστηρίζοντας και δημόσιε πολιτικές και μια κοινή στρατηγική. Σας άκουσα πολύ καλά. Ε, άκουσα πολύ καλά αυτά που είπατε κύριε Επίτροπε. Για την αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να επικεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας. Πρέπει να βοηθήσουμε τη βιομηχανία να εξάγει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο πιο ανοιχτό εμπορικό χώρο του πλανήτη και ταυτόχρονα οι επιχειρήσει μα να έχουν δυσκολίε στην πρόσβαση των αγορών τρίτων χωρών. Ολόκληρη η εμπορική μας πολιτική λοιπόν πρέπει να αναθεωρηθεί. Δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς στην υπόθεση αυτή. Και ελπίζω κύριε Επίτροπε ότι στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανίας αν καταφέρετε να το πετύχετε κάτι τέτοιο θα είναι πραγματικά ευχή έργο. Ευχαριστώ για τους ε, Σοσιαλιστέ και δημοκράτε, η κυρία Τόγια. Ε, ακόμα μια φορά μιλάμε για την βιομηχανία και για ανάγκη ανάκαμψη της ε, ε ευρωπαϊκής που πλήττεται από ε, μείωση της παραγωγής, ε, από ανεργία, από έλλειψη εξαγωγών κλπ. Ο, πρέπει κύριε Επίτροπε να κάνουμε μια κοινή μάχη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Χρειάζονται σημαντικά μέτρα. Ε, γίνονται, ε, γίνονται κατά χιλιάδες ε, οι απολύσεις χρειάζεται πραγματικά μια δράση ευρωπαϊκής διακυβέρνησης να αναλάβουμε τις ευθύνες μας πέρα από τα τυπικά με τη δημιουργία ενό διευθυντικού σώματος για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία που θα έχει μια εποπτεία όλων των ε, περιφερειακών ε, παραγόντων με στόχο την ανάπτυξη, με συμμετοχή και των τοπικών αρχών. Δεν μπορούμε να ε, παραμείνουμε αδρανείς απέναντι στην κρίση. Και χρειάζεται επίσης και η συνεργασία των τραπεζών, διότι συχνά ε, με το πρόσχημα ενός, ε, της έλλειψης ενός σαφού σε πλαίσιο αναφορά τα κεφάλαια φεύγουν έξω από την Ευρώπη. Η ανάκαμψη πρέπει να είναι εφικτή, διότι η Ευρώπη των 27 είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη ε, στην Ευρώπη κάποια στοιχεία αυτής της νέας στρατηγικής που αναφέρατε για την νέα βιομηχανική πολιτική ε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεγαλύτερη σύνδεση ανάμεσα στην παραγωγή και στις υπηρεσίες. Ε, το θέμα της ενέργειας και του κόστους και της εξάρτησης ενεργειακής. Αναφέρομαι επίσης τα μεγάλα προγράμματα ε, επενδύσεων για τις υποδομές, για τα αεροδρόμια που θα προσελκύσουν επενδύσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στρατηγικού χαρακτήρα. Επίσης αναφέρομαι στην έρευνα που είναι ε, κάτι το ε, προσιτό για μας. Επίσης την κατάρτιση, διότι θα πρέπει να υπάρχει ε, δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας, που είναι ένα μεγάλο ατού για την βιομηχανική πολιτική. Επίσης να μην, ξεχνάμε τον σύμμετρο ανταγωνισμό που δεχόμαστε από διάφορα διεθνή κέντρα. Ευχαριστώ ο, η κυρία Watson ο κύριος Watson για δύο λεπτά. Ευχαριστώ και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες που ε, δείχνουν το πραγματικό θάρρος ε, και προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτέ επιχειρήσει και να δίνουν δουλειά σε ανθρώπους. Η απουσία βιομηχανικής πολιτικής ή τουλάχιστον ε, ε, συνένεσης για την ανταγωνιστικότητα μέχρι στιγμής έχει εμποδίσει τις προσπάθειές του. Γι' αυτό οι φιλελεύθεροι καλωσορίζουν τα σημάδια μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής, το ότι εστιάζουμε στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου για να έχουμε πρόσβαση σε αγορές, ε, το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη για να δημιουργηθούν δίκτυα μεταφορών και ενέργειας και πληροφορικής, η επένδυση στην έρευνα και στην ε, καινοτομία, όπως η ανακοίνωση της προηγούμενης ε, εβδομάδας για το γραφένιο ή τη χατογράφηση του ανθρωπίνου εγκεφάλου και άλλα πράγματα. Καλωσορίζουμε επίσης τον ενεργειακό χάρτη για το 2050 και την εστίασή του σε φθηνότερη και καθαρότερη ενέργεια και την πράσινη ανάπτυξη. Όπως είπατε λοιπόν κύριε Επίτροπε θα πάτε στην Κρενόμπλ. Πείτε στους υπουργούς να μην επιτρέψουν στους ε, αρχηγούς των κυβερνήσεων να κόψουν από τους προϋπολογισμούς της έρευνας. Πρέπει να τους βάλετε στο μυαλό το τι μπορεί να επιτύχει η Ευρώπη εάν ενθαρρύνουμε την ευφυΐα των ελευθέρων ανθρώπων. Ε, φροντίστε λοιπόν να εστιάσετε στις επενδύσεις για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για τους πράσινους, ε, ο κύριος Λάμπερτς για δύο λεπτά. Συνάδελφοι, το δράμα αυτή τη στιγμή που ζει όλη η Ευρώπη από την ε, Φλωρεντία μέχρι τη Λιέγη έγινε σε μια παροχημένη βιομηχανία στην Ευρώπη. Γιατί κάνουμε ε, φορολογικά ε, δώρα ε, διότι κάθε φορά οι επιχειρήσεις παίζουν το χαρτί του εκβιασμού σχετικά με την με την κατάσταση. Τι κάναμε όμως, ανοίξαμε με ε, ανοίξαμε το, την Ευρώπη σε μια οικονομία του καζίνο όπου ε, μονά κερδίζω, ζυγά πληρώνει το κράτος. Και τελικά ε, θα πρέπει να δώσουμε βάρος στην πραγματική οικονομία ε, διότι υπάρχουν κέρδη που είναι ασύμβατα με μια ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία. Ε, η μεγάλη βιομηχανική όμιλη ε, είναι τα θύματα που πληρώνουν σήμερα. Τι πρέπει να κάνουμε όμως. Η απόλυτη προτεραιότητα είναι να κλείσουμε το δημοσιονομικό καζίνο το χρηματοοικονομικό καζίνο και να δώσουμε υποστήριξη στην πραγματική οικονομία. Ε, εκεί όπου κάποιοι ε, δείχνουν ε, να υποχωρούν, εμείς πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Επίσης πρέπει να περάσουμε στην οικολογική μεταμόρφωση της οικονομίας μας. Μέσω της πράσινης ενέργειας θα εξασφαλίσουμε τον καλύτερο τρόπο το μέλλον της βιομηχανίας μας. Και τέλος πρέπει να παραιτηθούμε από τη λογική των ελεύθερων συνολογών που αποσκοπεί μόνο στο εμπόριο ξεχνώντας περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κανόνες. Τη στιγμή που μιλάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένας ε, Ευρωπαίος στους τέσσερις βρίσκεται στο κατόφλι της φτώχεια. Αυτό ζητάει πραγματικά και επιγόντω αλλαγή πορείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάφτον για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στους τελευταίους τρεις μήνες του 2012 συρρυκνώθηκε 0,5% η οικονομία μας και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια τριπλή ύφεση που δεν έχει προηγούμενο στη δική μας σύγχρονη ιστορία. Σε όλη την περιοχή του ευρώ κανείς δεν θεωρεί ε, πως θα ε, έχει καλούς ρυθμούς ανάπτυξης φέτος. Η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε πως το ευρώ αποτελεί μια πλάνη ε, μια κακή σύλληψη που απέτυχε. Αποτελεί ένα ζουρλομανδία που περιορίζει τις δυνατότητες των λαών να αντιδράσουν. Είδαμε το μνημόνιο ε, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, η Κύπρος ακολουθεί και ποιος ξέρει και ποιος μετά. Για ποιο λόγο υπέρξε το ευρώ, για να έχουμε πιο στενή πολιτική ένωση, αλλά φέρνει να έχει φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και αναρωτιούνται όσοι βρίσκονται σε χώρες στην ανάπτυξη γιατί οι φόροι τους πηγαίνουν σε ε, ξένες οικονομίες που καταραίουν. Στη Γερμανία, την οποία γνωρίζω πολύ καλά, που θεωρούν όλοι τον βιομηχανικό τίγρη της Ευρώπης, δεν έχουμε ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης και δεν υπάρχει ε, ανάπτυξη. Ε, στέλνουν ε, όλοι τις θέσεις εργασίας στο εξωτερικό καταραίουν οι μικρομεσαίες. Εμείς στον Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουμε μια παρόμοια αλλά πολύ χειρότερη κατάσταση, πολύ ψηλή ανεργία και στους νέους ε, και βέβαια τα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη. Είναι μαύρο το μέλλον. Δεν θα έχουμε κάποια ανάκαμψη ή ανάταξη της βιομηχανίας. Στο παρελθόν ήμασταν γύρω στο 30% μερίδιο της βιομηχανίας στην οικονομία μας. Τώρα έχουμε πέσει στο 15-16%. Η ανάπτυξη ε, πνίγεται από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, στο σχιστολιστικό πετρέλαιο. Εκεί θα έπρεπε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ, ο κύριος Ενέν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήταν καιρό επιτέλου η Κομισιόν να ακούσει τη φωνή αυτών που εδώ στο Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια ζητούν μια πραγματική βιομηχανική πολιτική που να ανταποκρίνεται στι ανάγκε των πολιτών και των χωρών αντί, αντί ε, να παίρνουμε την αγορά σαν το μόνο κριτήριο. Ε, Αναγνωρίζουμε λοιπόν την προσπάθεια αυτή, αλλά περιμένουμε ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα, γιατί πολύ συχνά οι καλές προθέσεις της Κομισιόν σταματάνε εκεί που αρχίζουν τα συμφέροντα. Ναι, χρειάζεται μια πολιτική ε, διάσωσης και ανάπτυξης της βιομηχανική πολιτικής. Διαφορετικά, η Ευρώπη με την εξαίρεση της Γερμανίας και τον ορολάμων της ε, δεν θα είναι πια βιομηχανική περιοχή θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την καταστροφή αυτή την βιομηχανική. Ε, μεταξύ αυτών υπάρχει το κόστος της χρηματοδότησης και τα μέτρα λιτότητας. Ε, ε οι πολιτικές αυτές δεν χρηματοδοτούν τη βιομηχανία, αντίθετα την κάνουν να αιμορραγεί. Ε, η λιτότητα ε, οδηγεί σε ύφεση, σε κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης. Και το, οι, πωλήσει όπως στην αυτοκινητομηχανία ε, κατακυλάνε κατά 20%. Πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουμε ότι μια ε, επιχείρηση χρησιμεύει στο να παράγει ε, προϊόντα ε, χρήσιμα για το λαό μας και όχι να παχαίνει τους μετόχους της. Ευχαριστώ. Τελβώ για δύο λεπτά. Ήρθα, είδα, νίκησα. Αυτό κάνει η ArcelorMittal στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Έκλεισαν ε, το εργοστάσιο ε, στη Λιέγη. Και εγώ ζήτησα ε, και από το γραφείο το δικό σας και από αυτό το επίτροπο κύριο Αντόρ να δούμε εάν μπορεί να δημιουργηθεί ένας ιδρυκός πόλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δυνατότητες αναδιάρθρωσης. Αυτή η δράση επιτέλους ανακοινώθηκε για την Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία. Χαίρομαι. Όμως νομίζω ότι όπως και στην όπερα του Offenbach, όχι και στην περίπτωση με συγχωρείτε του εργασίου του Offenbach, φτάνει καθυστερημένο. 1.300 δουλειές θυσιάστηκαν έκτοτε. Αναρωτιέμαι λοιπόν για το πόσο ε, η εκτελεστική αρχή της Ευρώπης κατάφερε να αντιμετωπίσει τα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια χαλιβουργία. Τους εγκατέλειψε τους ανθρώπους αυτούς η αδύναμη Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να σπεύσουμε, να εξασφαλίσουμε στα κράτη-μέλη που ανησυχούν για το κλείσιμο αυτών των εργαστών των πώς θα τους δοθούν τα βιομηχανικά μέσα και εργαλεία για να εξασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας. Κάθε λύση που θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε ε, ε χαλιβουργία στην Ευρώπη υψηλή προστιθυμένη αξίας θα πρέπει να εξερευνηθεί χωρί ιδεολογικά κολλήματα. Καινοτομία, έρευνα για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Και επίση θα πρέπει να ζητήσετε από τι εθνικέ κυβερνήσει να χρησιμοποιήσουν όλη την πλειάδα εργαλείων που έχουν στη διάθεσή του, για να σώσουν τι χιλιάδε ατόμων των οποίων οι θέσει εργασία κινδυνεύουν. Όπω και στην αυτοκινητή βιομηχανία. Εδώ έχουμε πολυεθνικέ εταιρείε που πολύ συχνά ζυγίζουν από τη μία τα εργοστάσια και από την άλλη τους ανθρώπους με μοναδικό κριτήριο το κέρδος. Ευχαριστώ. Κυρίως Σενταρτέν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε ε, Επίτροπε, βρισκόμαστε σε μια στιγμή κλειδί. Οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη βρίσκονται σε σύγχυση, βρίσκονται σε απόγνωση, λιτότητα, απολύσεις, ενεργεία. Χρειάζεται δράση της Ευρώπης. Και με τη βιομηχανία υπάρχει εδώ μια μεγάλη ευκαιρία. Θα επικεντρωθώ στην ε, Χαλιβουργία λόγω της επικαιρότητα. Χρειάζονται δράσεις βραχυπρόθεσμες και στρατηγική, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Βραχυπρόθεσμα, σας ζητώ άμεσα πριν από τον Ιούνιο να παρουσιάσετε το σχέδιό σας για να δώσετε εμπιστοσύνη στους ε, ε, επενδυτές θα πρέπει να ακούσετε τους ε, ε, υπουργούς βιομηχανίας και κυρίως τον Βέλγο για να ε, διατηρηθεί η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Με τους συναδέλφους σας του ανταγωνισμού θα πρέπει να, κάνετε, να προτείνετε μέτρα ούτω ώστε το δημόσιο ή οι ιδιώτες να, προωθηθούν, να, να παρατηρηθούν να επενδύσουν. Χρειάζονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία να ξαναποκτήσει το ρόλο της. Ε, διότι θα πρέπει αυτή να είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Πέραν αυτού, βιομηχανική πολιτική για τους ε, ε, τομείς που υφίστανται αλλαγέ, χρειάζεται, για να γίνει αυτό, χρειάζεται ένα πυλώνα, όπω υπάρχει στα πλαίσια τη γεωργική ή τη αλληλευτική πολιτική. Μεσοπρόθεσμα τέλο, η πολιτική θα πρέπει να περνάει μέσα από ε, επενδύσει ε, μέσα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, καθώ επίση και ε, με θεωρήσει ε, ε περιβαλλοντικέ και κοινωνικές. Και, ε, εν πάση περιπτώσει, θα σταματήσουμε αυτό το ε, βιομηχανικό ντάμπινγκ. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Τζιρόν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ρωτώ. Σήμερα ποιος είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος που είναι υπεύθυνο για τη Χαλιβουργία. Δεν είναι ο κύριος Τατζάνη. Είναι ο κύριος Μιτάλ. Αυτός είναι ο κύριος που εδώ και χρόνια είναι ο εκπρόσωπος της σιδηροβιομηχανίας στην Ευρώπη που έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου και που επιτρέπει στους μέσα την αναδιάρθρωση, στους άλλους όχι, ε, φέρνοντας αντιμέτωπους περιοχές και κράτη ε, στην Ευρώπη ε, που λέει σε όλους ότι θα πρέπει να σφιχτούν. Δηλαδή να σφιχτούν γιατί, να περιμένουν ποιος είναι ο επόμενος που θα πέσει. Νομίζω πως είναι δική σας ευθύνη σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, καλείται να μας εγγυηθεί μια πραγματική βιομηχανική και χαλβουργική πολιτική να αποφασίσει και να θέσει εφαρμογή. Από το 2009 μας λέτε πως ναι βρίσκεται στα σκαριά. Είμαστε το 2013 και μας ανακοινώνεται ένα σχέδιο δράσης για τον Ιούνιο του 2013. Μα παραδεχτείτε το, υπάρχουν λόγια ανησυχία και σας λέω γιατί πρέπει γρήγορα εσείς να δείτε τα θέματα που δεν είναι μόνο τα περιβαλλοντικά ή τις απαιτήσει που ε, επιβαρύνουν τη χαλιβουργία. Όχι. Ο μόνος τρόπος είναι η ανάταξη, η πράσινη ανάκαμψη. Έτσι μόνο θα σώσετε τη χαλιβουργία. Δεύτερον, θα πρέπει να ελέγξετε και να, να επαληθεύσετε αν οι κανόνε ανταγωνισμού σε κάθε περίπτωση έγιναν σεβαστέ. Γιατί νομίζω ότι στο χάλιβα εκεί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Τρίτον, θα πρέπει να προστατεύσουμε την τεχνολογία μα, την καινοτόμο, με τελωνιακού δεσμού, με, εξαγωγικού, με ε, ε, περιβαλλοντολογικούς δεσμούς κτλ. Γρήγορα θα πρέπει να εργαστείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, ο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πλήττεται, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, αλλά οπωσδήποτε βλέπουμε πως τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης ε, φτάνουν πέρα από την ευρωπαϊκή οικονομία. Δυστυχώς, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάμε μόνο για απορρίθμιση και για το να μην εμποδίζουμε με τις ε, ρυθμίσεις την ελεύθερη αγορά. Αλλά αντί να κάνουμε κάτι, μόνο λόγια έχουμε, οι ρυθμίσεις αυξάνονται, όλο και περισσότερο, αυξάνονται, και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό και Έχουμε και το πακέτο του κλίματος ε, και μετά μας προξενεί κατάπληξη το ότι κάποιος άνθρωπος θέλει να πάρει τη χαλιβουργία του και να φύγει. Μα ο άνθρωπος ξέρει και μετράει τα κέρδη του. Βλέπει τι τον ε, συμφέρει και αν τον συμφέρει να συνεχίσει να παράγει στην Ευρώπη. Εάν συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας που ανεβαίνουν λόγω του πακέτου του κλίματος. Κάτι το οποίο αναπόφευκτα οδηγεί σε υψηλότερη τιμή ενέργειας. Άρα υψηλότερο κόστος παραγωγής του χάλιβα. Οπότε ο επιχειρηματίας θα πάει αλλού την παραγωγή του. Γιατί επιχειρηματίας είναι, δεν κάνει φιλανθρωπία. Δυστυχώ αυτό είναι αποτέλεσμα και τη δική μα δραστηριότητα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη το ότι το πακέτο του κλίματο απορρίπτεται από τι ΗΠΑ, στη Βραζιλία, την Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να είναι πρωτοπόρο σε αυτόν τον τομέα αλλά δρά ει βάρο της ίδιας της, της οικονομίας. Ε, πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ε, πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να στηρίξουμε την οικονομία μας. Είμαστε σε κρίση. Πρέπει να μειωθεί το ενεργειακό κόστος, να ξανασκεφτούμε το κλιματικό αυτό πακέτο γιατί θα επηρεάσει την κατάσταση στην Ευρώπη με το να μειώσει τον αριθμό ε, θέσεων εργασία ε, στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θέλουμε να πληρώσουμε ένα τέτοιο τίμημα. E Ευχαριστώ, κυρία Καρβάλο, για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, η στρατηγική για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική που θα βασίσει στην καινοτομία, στην αποδοτικότητα σε επίπεδο κόστος και στην ορθή χρήση των ανθρωπίνων πόρων. Καινοτομία, ουσιαστικό συστατικό γιατί δεν μπορούμε να αρθρώσουμε μια σωστή βιομηχανική πολιτική αν δεν βασίζεται αυτή στην καινοτομία και στην αποδοτικότητα σε φυσικές, ε, στις πρώτες ύλες και κυρίως στην ενέργεια δηλαδή βιώσιμη ανάπτυξη και βιομηχανική ανάπτυξη. Θα πρέπει να βασιστούμε στις δυνατότητές μας για να καινοτομήσουμε μέσω της κατάρτισης, της παιδείας, αυξάνοντας τον αριθμό των επιστημόνων σε τέτοιους κλάδους όπως και τον αριθμό των μηχανικών στην Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφερθώ στην εκ νέου βιομηχάνηση της Ευρώπης. Το πρώτο είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία πριν ε, το Συμβούλιο Βιομηχανίας ε, Ανταγωνιστικότητας, με συγχωρείτε, τον Δεκέμβριο. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Έτσι θα έχουμε μόνο ένα μοχλό που θα φέρει την ανάπτυξη. Ελπίζουμε πως ο προπολογισμός 2014-2020 θα στείλει ένα σημαντικό μήνυμα που θα δώσει προτεραιότητα στις πολιτικές που περισσότερο συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην εκπαίδευση και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντρές για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα πρέπει να ε, επενδύσουμε στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας μια ανάπτυξη και να δώσουμε μια απόκριση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Σήμερα βλέπουμε ποιες είναι οι δυσκολίες. Έχει πάρα πολλές γιατί είμαστε σε μια περίοδο, ε, τη χαμηλότερη περίοδο επενδύσεων στη βιομηχανική πολιτική τα τελευταία δέκα χρόνια. Κλείνουν ε, μερικά ή πλήρως εργοστάσια και ε, εμοραγούν οι θέσεις εργασίας και έχουμε πρόσφατες ε, περιπτώσεις στη Γάνδη για παράδειγμα, στη Λιέγη, ε, στην ε, Ισπανική Χαλιβουργία, στην περιφέρεια Αστούριας αντιμετωπίζουν σημαντικότητα προβλήματα. Ακόμα όμως είμαστε στην αιχμή του δόρατος και θα πρέπει να παραμείνουμε με μια πολιτική αυτοματοποίησης παραγωγής και με προσπάθειες και στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη φαρμακοβιομηχανία και στην αεροναυπηγική και στην αυπηγική. Θα πρέπει να δούμε ποια θα τα μέτρα προτεραιότητας για την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα από τις περιφέρειες στα κράτη και από εκεί στην Ευρώπη και το αντίστροφο, καλύτερη διαχείριση, καλύτερη κανόνες, όχι εθνικές λύσεις που μας αποδημονούν και μας κατακαιρματίζουν. Σας ζητούμε λοιπόν κάποιες δράσεις για να λειτουργήσει η ενιαία αγορά, να λάβουμε υπόψη όλη την αλυσίδα τιμών των ε, προϊόντων από τις πρώτες ύλες μέχρι τις υπηρεσίες και κάποια εγκάρσια μέτρα, να δούμε ποιο είναι το ενεργειακό μοντέλο που μας λείπει και επίσης πρόσβαση στα δάνεια. Τι θα γίνει με το Horizon 2020 και σας απευθύνω μία έκκληση. Πείστε το Συμβούλιο, πείστε τους Υπουργούς Βιομηχανίας και Επιστημών των διαφόρων κρατών μελών πώς η βιομηχανία μπορεί να φέρει τη λύση σε αυτή την κρίση. Ευχαριστώ ο κύριος Λάγκε για ένα μισή λεπτό. Ehm, Μάλιστα, δεν είναι εδώ οι, ομιλητές αυτοί, άρα αρχίζουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Ο πρώτος, ομιλητής είναι ο κύριος Λούαν. Ευχαριστώ. Η διεθνής μας ανταγωνιστικότητα βασίζεται στην ε, βιομηχανία. Χωρίς ε, βιομηχανία δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο σημαντικό ρόλο. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε κάποια μέτρα δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους νέους ε, mm για να καλύψουμε τις ανάγκες της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας. Ε, χρειαζόμαστε ορισμένα προγράμματα για τεχνολογική εκπαίδευση των νέων για να έχουν την δυνατότητα να εξειδικευτούν και να δουλέψουν σε άλλα κράτη-μέλη. Και τέλος πρέπει να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα των νέων και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια και αυτό σε όλα τα κρατη Ευχαριστώ. Μπαζέσκου. Κυρία Μπαζέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζούμε σε μια εποχή που η έλλειψη βεβαιότητας, η έλλειψη χρηματοδότησης ε, εμποδίζουν τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα για να διορθώσουν την οικονομική κατάσταση. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να κάνει τη νέα βιομηχανική επανάσταση, να κάνει την Ευρώπη ένα μέρος ελκυστικό και πάλι για τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές. Μια νέα βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να βασιστεί σε νέες μεθόδους παραγωγής, σε καινοτόμα υλικά και σε έξυπνα συστήματα επικοινωνίας. Η ρουμανική βιομηχανία έχει και αυτή ε, υποστεί ε, ύφεση και παρακμή. Πιστεύω ότι η βάση οποιασδήποτε ε, ανάκαμψης ε, βρίσκεται σε τομείς όπως είναι ε, τα ορυχεία και το φυσικό αέριο. Ε, τα χρυσορυχεία, παραδείγματο χάρη, είναι μια καλή ευκαιρία να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και Επίσης, η παραγωγή φυσικού αερίου θα μπορούσε να δημιουργήσει απασχόληση και να μας δώσει και ενεργειακή ανεξαρτησία. Ευχαριστώ. Ο κύριος, η κυρία Μαστάρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγετική οικονομική δύναμη στον πλανήτη. Αυτό βέβαια δεν το είδαμε τα τελευταία χρόνια. Αιτία γι' αυτό είναι η έλλειψη, όπως είπαμε, βιομηχανικής ε, πολιτικής. Έχουμε το πρόγραμμα για την καινοτομία 2020, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Σταγιάννη για τη μυρία θέσεων εργασίας. Ε, πρέπει να συμβιβαστεί επίσης και με την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Οι μεγάλες βιομηχανίες στον κόσμο κινητοποιούνται και είναι προσανατολισμένες προ την ε, τεχνολογία. Εμεί είμαστε προσανατολισμένοι προ το περιβάλλον. Αυτό κοστίζει, ειδικά σε καιρό κρίση. Εδώ πέρα πρέπει να βρούμε έναν συμβιβασμό, γιατί οι ανταγωνιστέ μα δεν κολλάνε σε δικαιώματα εκπομπών και τέτοια πράγματα, τα οποία εμάς μας εμποδίζουν στην ανταγωνιστικότητα. Σας ευχαριστώ. Πρέντεργκάστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά μπορούμε να πούμε για την έλλειψη συντονισμένων βιομηχανικών πολιτικών της ε, τελευταίας δεκαετία. Εμπιστευόμαστε πάρα πολύ τι ε, αγορές ε, οι οποίες ε, κοιτάνε μόνο τα βραχυπρόθεσμα κέρδη και τα αποτελέσματα τα ξέρουμε. Σήμερα όμως θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο ποια είναι η απόψή του για συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να μην διαβρωθεί άλλο η βιομηχανική μας βάση και να ανακτήσουμε θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη παρέχει νομική προστασία στα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που προερχόνται από συγκεκριμένες περιοχές. Θα ήθελα να προτείνω η προστασία αυτή να επεκταθεί και σε ε, βιομηχανικά αγαθά, όπως παραδείγματο χάρη το κρίσταλο του Waterford, πολύ γνωστό προϊόν υψηλής ε, ποιότητας και χειροτεχνίας ε, στην Ιρλανδία. Όταν έκλεισε η βιομηχανία το 2009 και χάθηκαν 600 εργασίες, η εταιρεία η οποία απέκτησε την εταιρεία μετέφερε την παραγωγή στο εξωτερικό, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το όνομα κρίσταλο του Waterford, μια παράδοση δηλαδή αιώνων. Οπωσδήποτε θα πρέπει προς το συμφέρον και των εργαζόμενων ε, και των υπολείπων να υπάρξει ένα σύστημα γεωγραφικής προέλευσης για κάποια βιομηχανικά αγαθά. Ευχαριστώ. Ονορεύολε Ταραμπέλα. κύριος ε, Όντω η χαλιβουργία αξίζει μια συζήτηση από μόνη της γιατί είναι στην επικαιρότητα. Από το 2008 30% της ευρωπαϊκής παραγωγής ε, η ευρωπαϊκή μάλλον παραγωγή μειώθηκε κατά 30% και βλέπουμε μια μετεγκατάσταση της παραγωγής. Μιλήσατε για μια βιομηχανία σύγχρονη και πράσινη. Είναι γεγονός ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία έκανε την προσπάθειά της. Αλλά η βιομηχανή... Ε, έχουν πιο μακροπρόθεσμη εικόνα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν πάρουμε τον, ε, την, ε, τον Λάξι Μιτάλ στη Λιάγη αλλά και αλλού, στην Ρουμανία και στη Γαλλία, πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν κάστες. Ε, υπάρχουν ε, πολίτες με ίδια δικαιώματα που αξίζουν όλοι τον ίδιο σεβασμό. Και άρα, σε σχέση με αυτό, όπω είπε ο κ. Επίτροπε, βλέπουμε μετακατάσταση εκτό τη Ευρώπη και γι' αυτό βασιζόμαστε σε εσά και στου συναδέλφου σα, στους συνάδελφό σα για το εξωτερικό εμπόριο, ώστε να ληφθούν διαρθρωτικά μέτρα ε, και για τι ε, ε, κρατικέ ενισχύσει, παραδείγματο χάρη, αλλά και ε, θα πρέπει ε, τα εργαλεία αυτά να μην ε, τα παραχωρούμε σε άλλους και εμείς να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Κυρία Γιανακοδάκη, ήθελα να σχολιάσω την ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης. Η Κάιλ έχει η βιομηχανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο προσέφερε γύρω στις 450 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την τελευταία τέτοια βιομηχανία στην ε, Ευρώπη. Βρίσκεται στην περιφέρειά μου στο Λονδίνο. Έχει απολύσει 28 άτομα. Είχε ε, χασούρα 28 εκατομμυρίων ευρώ και ε, άλλα 50 άτομα δουλεύουν με μειωμένο ωράριο τη στιγμή που οι τιμές της ζάχαρης στην Ευρώπη είναι 80% πάνω από τις παγκόσμιες τιμές. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρόσβαση στις αυτό μπορεί να το κάνει η Κομισιόν. Η Κομισιόν μπορεί να προστατεύσει θέσει εργασία και να σώσει μία από τις παλαιότερες βιομηχανίες της Ευρώπης, αλλά αρνείται αυτή τη στιγμή να δώσει μια χείρα βοηθεία παλαιότερε ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο. Θα πρέπει το ζαχαροκάλαμο, η εισαγωγή του δηλαδή, να δωσει μια χειρα βοηθεια στην βιομηχανια Ζάχαρη απο ζαχαροκαλαμο θα πρεπει το ζαχαροκαλαμο η εισαγωγη του δηλαδη να συμπεριληφθει για να μειωθεί και το κόστος της ζάχαρης και να βοηθήσει ε, αυτό τον κλάδο διασφαλίζοντας ε, ίσους όρους ανταγωνισμού με τους παραγωγούς από ζαχαρότευτλα. Ευχαριστώ. Ονορεύολε Τζούμπερ. Τζούμπερ. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, στην Πορτογαλία καταστρέφονται χιλιάδες ε, θέσεις εργασίας και αυτό κάνει τη χώρα μας να εξαρτάται περισσότερο από ό,τι ποτέ από τον εξωτερικό κόσμο από τον έξω κόσμο. Έχουμε χάσει τόσες πολλές ε, θέσεις εργασίας και τόσες πολλές επιχειρήσεις έφυγαν από τη χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια. Πιστεύω ότι η κατάσταση είναι παρόμοια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρόλο που στην Πορτογαλία είναι πολύ χειρότερη. Ε, ο βαθμός αποβιομηχάνησης στην Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ ε, μεγαλύτερος από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, βιομηχανικό κεφάλαιο εγκατέλειψε την Πορτογαλία και έτσι δεν αξιοποιείται πλήρως το δυναμικό της χώρας, μιας περιφερειακής χώρας της Ευρώπης. Ε, ο μόνος τρόπος να, επανέλθει η βιομηχανική ανάκαμψη στην Πορτογαλία είναι μέσω δημόσιων επενδύσεων. Αυτό είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις δημόσιες επενδύσεις από τη βιομηχανία, από τις εθνικές κυβερνήσεις. Διαφορετικά δεν πρόκειται να έχουμε βιομηχανική ανάκαμψη στην ε, Ευρώπη. Ο κύριος Πάσκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, η ευρωπαϊκή οικονομία μένει στάσιμη. Οι επιχειρήσεις κλείνουν ε, μαζικές απολύσεις και όσο μεγαλώνει η ανεργία τόσο περισσότερο επιβαρύνονται τα κρατικά ταμεία. Και υπάρχουν όμως και ισχυρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εγγράφουν κέρδη και μάλιστα παγκοσμίω οικοδομούν οι εργοστάσια. Η Volkswagen στην Κίνα, η Fiat στη Βραζιλία λοιπά. Και έτσι δίνουν ε, δουλειά σε Κινέζους, Ρώσους κτλ. Δουλειά που θα μπορούσε να γίνει εδώ πέρα. Αν λοιπόν θέλουμε να αναβιώσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, ακριβώς πρέπει να ζητήσουμε από αυτές τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις ε, να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί κλείνουν εδώ τα εργοστάσια και τα ανοίγουν αλλού στο παρελθόν ε, ο πλούτος Ευρώπης ε, δημιουργούταν εδώ πέρα και μετά γινόταν εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ στο... Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Μιλάμε για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως στη Βουλγαρία η βιομηχανία καταστράφηκε προ-κρίσης. Τρεις κυβερνήσεις φρόντισαν γι' αυτό. Μία κέντρο δεξιά, μία κέντρο μια κέντρο αριστερή έκαναν κάθε προσπάθεια για να συμβεί αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση κοίταζε και ενίσχυε αυτές τις κυβερνήσεις και όπως είπε και η κυρία Γιανακουδάκη για το τι συμβαίνει στη ζάχαρη και για την απειλή ε, της συγκεκριμένης βιομηχανίας θα μπορούσα και εγώ να πω το ίδιο για την Βουλγαρία Γι' αυτό υπάρχουν και πολλοί ε, Βούλγαροι οι οποίοι δεν θένε πλέον να ανήκουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, μια πολιτική παρατήρηση. Μετά από πολλά χρόνια η Ευρώπη ξανά ε, θέτει την έμφαση της, ε, θέτει την έμφαση στα πλαίσια της οικονομίας της στην πραγματική οικονομία. Μετά από αρκετά τέρμινα που όλη η προσοχή ήταν επικεντρωμένη στις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες γενικότερα, με την έναρξη της δεύτερης θητείας του Μπαρόζο άλλαξε μια τάση τέτοια και ξαναρχίσαμε να μιλάμε για την βιομηχανική πολιτική. Σε 15 χρόνια κοινοβουλευτικής ε, δραστηριότητας, εγώ ανάμεσα στο 1994 και το 2008 συμμετείχα σε πολλές συζητήσεις για την βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη. Για το πρόβλημα του ποια βιομηχανική πολιτική πρέπει να έχουμε. Και θα έλεγα μάλιστα και στο επίπεδο του Συμβουλίου ε, πάντοτε πολύ λίγος λόγος έγινε, γινότανε για την βιομηχανική πολιτική. Και τελικά έγινα ο αρμόδιος επίτροπος. Θυμάστε ότι ο επίτροπος Δαβινιών είχε ε, ε, ένα σχέδιο για τη βιομηχανική πολιτική. Ακόμα και οι αρμοδιότητες που δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιομηχανική πολιτική είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Όμως ε, χρειάζεται μια επιλογή υπήρξε μια, πολιτι... μια απόφαση πολιτικού τύπου που μας ε, έκανε να επικεντρωθούμε πάλι στις επιχειρήσεις, στη βιομηχανία για να καταπολεμήσουμε την κρίση. Γιατί αν είχαμε μια οικονομία που βασίζεται μόνο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, απλώς ε, γυρνάει το χρήμα και καταλήγει σε συγκεκριμένες τσέπες. Η βιομηχανική πολιτική, η πολιτική των επιχειρήσεων δημιουργεί νέο πλούτο και πάνω απ' όλα επιτρέπει η αναδιανομή αυτού του πλούτου χρησιμοποιώντας την αγορά όχι ως ε, αυτό σκοπό αλλά ως μέσο για να ε, υλοποιηθεί η κοινωνική πολιτική. Έγινε αυτή η αλλαγή και δεν ήταν τυχαίο και δεν ήταν ούτε εύκολο. Κυρία Ντουράν, το να πείσουμε ολόκληρη την Επιτροπή ότι υπάρχει ένας στόχος που πρέπει να επιτύχουμε μέχρι το 2020 σε αυτούς που έχουμε να προσθέσουμε ένα ακόμα στόχο δηλαδή ότι το 20% του ΑΕΠ θα πρέπει να είναι καρπός της ε, βιομηχανικής παραγωγής μέχρι το 2020. Είναι μια πολιτική επιλογή τεράστια σημασίας. Και επίσης και ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, χαιρέτησαν αυτό το νέο στόχο. Το να περάσουμε τώρα σε συγκεκριμένη υλοποίηση από τα λόγια αυτού του στόχου δεν είναι κάτι εύκολο. Γιατί μια αλλαγή πολιτική ε, πρέπει να έχει πρακτικές συνέπειες που απαιτούν και κάποιο χρόνο. Έδειξα, έδωσα ε, μεγάλη προσοχή στον κύριο Μιτάλ και συνολικά στην κατάσταση της ε, χαλιβουργίας που αφορά και την πατρίδα μου. Ε, μην ξεχνάμε τη χαλιβουργία του Τέρμη. Δώσαμε ζωή σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Πριν από τις καλοκαίρες διακοπές του 2012. Ε, μια συνεδρίαση όπου ήρθαν συνδικαλιστές ε, από όλες τις βιομηχανίες, τις τόσες πολλές στην Ευρώπη του κυρίου Μιτάλ. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η ομάδα όπου συμμετείχε όχι μόνο η βιομηχανία, όχι μόνο οι συνδικαλιστές αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι αποτελεί πλήρες μέλος αυτής της ομάδας εργασίας καθώς επίσης και η πρόεδρος Περβάν Σπερές και ε, ο πρόεδρος Σαρτόρη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε πλήρως λοιπόν σε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου που χρειάζεται και αυτή χρόνο βεβαίως ε, για να βρει λύσεις. Στις 12 του μήνα θα συμμετάσχει και ο, ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για θέματα απασχόλησης. Ο Επίτροπος Νταβνιών ε, είχε ένα σχέδιο για την Μιχαηλυπουργία. Ε, αυτό είναι το ε, μοντέλο για μας. Ε, στις 12 του μήνα, εκτό από του συνδικαλιστέ, εκτό από του βιομηχανού μεταξύ των οποίων ο κ. Μιτάλ, εκτό και από του εκπροσώπους του Βρεγού Κοινοβουλίου και τον Επίτροπο κύριο Άντορ, ε, θα είναι στι Βρυξέλλες και οι Βέλγοι οι υπουργοί που, θα είναι υπεύθυνοι, που είναι υπεύθυνοι για τη βιομηχανική πολιτική θα είναι και ο Γάλλος υπουργός και όλα τα κράτη-μέλη με συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα προσπαθήσω να συντονίσω όλα αυτά και να βρω ε, λύσεις ώστε να αποφύγω συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών. Το ίδιο συμβαίνει και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν είναι ομοιογενείς όλες οι θέσεις ε, της ε, ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, αποφύγουμε τη σύγκρουση εντός του κλάδου. Υπάρχει πάντοτε το πρόβλημα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι ε, στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών. Η επιλογή αυτή όμως σημαίνει και θυσίες. Εγώ το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορούμε ε, όταν ε, δεν υπάρχει μια παγκόσμια συμφωνία να πάμε πάνω από το στόχο του 20% της μείωσης γιατί η βιομηχανία μας δεν είναι σε θέση να ξεπεράσει αυτό το στόχο. Έστω και θα ήταν ευκταίο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν θέλουμε να εμποδίσουμε βέβαια την μετεκατάσταση που είναι τεράστια ζημιά ε, και για τους στόχους μας όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Γιατί η βιομηχανία, η βιομηχανία πάει να παράγει εκεί όπου δεν υπάρχουν κανόνες, ε, ισχυροί κανόνες κατά των κλιματικών αλλαγών. Άρα αυτό είναι εις βάρος και της δράσης μας υπέρ του περιβάλλοντος. Και όσον αφορά την χαλιβουργία, για συγκεκριμένα τώρα πράγματα, γιατί δεν κάνουμε μόνο γενικές ε, πολιτικές επιλογές, έχουμε ε, εντάξει την χαλιβουργία και όσον αφορά ε, τις ποσοστώσεις ε, με ενισχύσεις του κράτους μέχρι το 80% μεταξύ των κλάδων που ε, επιτρέπεται η κρατική ενίσχυση. Και αυτό ήταν μια επιλογή που οι ίδιοι οι συνδικαλιστές αναγνώρισαν σαν πολύ αξιέπαινη επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποια πράγματα λοιπόν έγιναν ήδη. Πριν από την ε, υλοποίηση του σχεδίου δράση που απαιτεί, όπως σας είπα, κάποιο χρόνο γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να βρεθούν ε, οι συμφωνίες, να καταλήξουμε σε συμφωνίες και να ε, εγκριθούν αυτά από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Παρακολουθούμε όμω με μεγάλη ε, προσοχή και ο κύριος Σαλμούνια εξάλλου που είναι υπεύθυνο για την πολιτική ανταγωνισμού. Παρακολουθούμε με κάθε προσοχή την ε, υπόθεση αυτή της αγοροπολισίας που όπως είπε η πρόεδρος Αντζελίλη αφορά μια σημαντική φιλανδική εταιρεία που έχει να κάνει με ε, θέματα ανταγωνισμού γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι κανόνες της ε, βιομηχανικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της πολιτικής ανταγωνισμού που μας οδηγούν σε, αλλαγή, σε επιλογές που ε, μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις, να έχουν συνέπειες που απαιτούν ε, στη συνέχεια νέες παρεμβάσεις. Εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν ε, εργάζεται σωστά και όσον αφορά την προστασία των επιχειρήσεών μας. Δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε ένα σεμινάριο που ήταν αφιερωμένο ακριβώς στην ανταγωνιστικότητα του ε, βιομηχανικού μας συστήματος που θέλησε να πραγματοποιηθεί ο, ε, πρόεδρος Παρόζο και βεβαίως ε, όλα αυτά σχετίζονται και με την ε, εμπορική πολιτική μας. Δεν μπορούμε να έχουμε μια αφελή πολιτική ε, για το εμπόριο. Μέτρα αντι-dumping που ακριβώς υιοθετήθηκαν για να μην υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό. Είμαι απόλυτα ε, όσον αφορά το level playing field. Ε, φυσικά πρέπει να υπάρχει παγκόσμιο ανταγωνισμός, αλλά για το παιχνίδι πρέπει να ισχύουν πάντα οι ίδιοι κανόνες. Δεν μπορούμε να παίζουμε το, το ίδιο παιχνίδι στις Βρυξέλλες 11 ε, εναντίον 11 και μετά να πάμε στο Πεκίνο να παίζουμε 9 εναντίον 13 γιατί είναι χαμένο από χέρι το παιχνίδι αυτό και υπάρχουν πολλά προβλήματα και όσον αφορά την προστασία του ε, know-how μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ε, να εφαρμόζουμε έναν προστατευτισμό αλλά θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε τις ικανότητές μας όπως επίσης εργαζόμαστε και για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας στον τομέα της ε, ε, τεχνολογίας εχμής. Στις 12 του μήνα στην Γκρενόμπλ θα γίνει μια συνάντηση με τους ε, υπουργούς κάποιων χωρών στο κέντρο της Γκρενόμπλ, χωρών που είναι οι πιο ανταγωνιστικές όσον αφορά ε, τις τεχνολογίες αυτές. Και όσον αφορά τον ορίζοντα του 2020, αυτή είναι μια επιλογή που περιλαμβάνει μια, επιλογή που περιλαμβάνει μια αλλαγή. Για πρώτη φορά η έρευνα δεν θα είναι αυτός σκοπός, αλλά θα αποσκοπεί ε, και θα αποβλέπει προς την ε, βιομηχανική πολιτική, διότι δεν μπορούμε πια να δεχόμαστε οι κίνεζικοί ή οι άλλες βιομηχανίες να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της δικιάς μας έρευνας ε, για, για τον λόγο αυτό χρειάζεται στενή σχέση ανάμεσα στην έρευνα, το πανεπιστήμιο και τις επιχειρήσεις. τέτοια λάθη δεν μπορούμε πια να επιτρέψουμε στον εαυτό μας. Δεν είναι δευτερεύον πλέον αυτό το θέμα. Η επιλογή της ε, Κομισιόν ήταν πάρα πολύ σαφής όσον αφορά αυτό το σημείο. Και η πολιτική ε, για την εκ νέου εκβιομηχάνηση της Ευρώπης ε, περιλαμβάνει και αυτή τη διάσταση κατά της μετεκατάστασης αλλά υπέρ της διεθνοποίησης της βιομηχανίας. Ε, όταν δεκάδες ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πάνε και κάνουν τις δραστηριότητές τους ε, στην Νότια Αμερική και σε όλα τα σημεία του κόσμου. Χρειαζόμαστε μια βιομηχανική πολιτική σύγχρονη, υπεύθυνη, με σεβασμό προς το περιβάλλον. Πρόκειται για μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση ε, φυσικά ε, σας είπα ότι χρειάζεται χρόνος, δεν λείπουν και οι αντιδράσεις και δεν θα λείψουν και στο μέλλον. Ε, η εργασία ε, της ομάδας υψηλού επίπεδου έδωσε σαν αποτέλεσμα μια άλλη ομάδα εργασίας που ασχολείται με την αυτοκινητοβιχανία που πάσχει σήμερα, όπως και η χαλιβουργία. Κάνουμε πολλά πράγματα και για αυτό τον κλάδο, με αποτελέσματα ε, που αναγνώρισαν οι επιχειρηματίες. Ε, επίσης μιλάμε ε, για τα ναυπηγεία με προσπάθειες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες για να αποκτήσει η Ευρώπη μια νέα σύγχρονη βιομηχανική πολιτική. Πρέπει να πάω και να πω ε, στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει να μετατραπεί το Συμβούλιο σε Συμβούλιο Βιομηχανίας και Ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να τα συζητάμε αυτά ξεχωριστά σε δύο ή τρία ε, συμβούλια. Όταν πρόκειται ε, για πολιτικές αποφάσεις πρέπει να είναι παρόντες οι υπουργοί. Αυτό είναι απαραίτητο. Γι' αυτό ε, για πρώτη φορά άτυπα θα συγκαλέσω όλους τους υπουργούς για να μιλήσουμε για την κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε όλους τους άλλους κλάδους. Ε, το γράμμα που έλαβα πριν από μερικούς μήνες από 7 ε, Ευρωπαίους Υπουργούς Βιομηχανίας που ζητούσαν μια ισχυρή δράση εκ μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δράση συντονισμού, ήταν ένα μήνυμα το οποίο ε, εισέπραξα και το μετέτρεψα σε συγκεκριμένη δράση. Επαναλαμβάνω, οι αρμοδιότητες που έχουμε είναι αυτές που είναι και αυτές που προβλέπονται από τη συνθήκη. Επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά δεν ήταν αυτές που είχε ο Επίτροπος Νταβινιόν όταν χάραξε το πλάνο για την Χαλιβουργία. Το είπε ίδιος. Αν είχα τέτοιε ε, εξουσίες σίγουρα θα είχα κάνει μια πρόταση ε, προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχω την εξουσία, δεν έχω την αρμοδιότητα όμως να το κάνω και πρέπει να σεβαστώ τη συνθήκη. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να διαβεβαιώσω όλους τους ευρωβουλευτέ που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και είναι καλό που έγινε αυτή η συζήτηση για τη βιομηχανική πολιτική, γιατί αυτό είναι ένδειξη μια αλλαγή. Α συνεχίσουμε να συζητάμε τι ιδέε, τι προτάσει το πώς θέλουμε να είναι μια ε, σύγχρονη ε, βιομηχανική πολιτική που να σέβεται στο περιβάλλον, που να είναι πράσινη η οικονομία, που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Δεν μπορούμε ε, βεβαίως να σκεφτούμε ότι θα ανταγωνιστούμε ε, όσον αφορά την ποσότητα με χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, οι χώρες της Νότιας Αμερικής. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε όμως την ποιότητα. Και σε αυτό μπορούμε να έχουμε ακόμα πολλά ατού για να κερδίσουμε αυτή την πρόκληση. Σκεφτείτε όλες τις συνέπειες, όλες τις επιπτώσεις που θα έχουμε χάρη ε, στο δορυφορικό μας ε, πρόγραμμα Γαλιλαίο και ε, τις στο διάστημα. Η ίδια η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου οργάνωσε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη ακριβώς στις υπηρεσίες και στις ε, επιχειρήσεις ε, υπηρεσιών που θα χρησιμοποιήσουν επί της γης ε, τα σήματα του Γαλιλαίου για τη γεωργία, για τις μεταφορές, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό είναι το βιομηχανικό μοντέλο που έχουμε στο μυαλό μας. Ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία που συχνά έχει επιφυλάξεις για κάποιες επιλογές ε, των κοινοτικών πολιτικών. Όταν πρόκειται για μια τέτοια ε, μοντέρνα βιομηχανική πολιτική, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να έχουμε το θάρρος και την δύναμη να συνεχίσουμε, να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο που έχουμε χαράξει, να συνεχίσουμε να ε, ενισχύουμε τις αλλαγές και εγώ έχω το καθήκον να κάνω ό,τι μου είναι δυνατόν, αλλά χρειάζομαι την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσω να ε, επιτύχω αυτή την αλλαγή πορείας που θέλησε ο, ο ίδιος ο πρόεδρος Μπαρόζο με την σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν. Οι επιλογές έχουν γίνει πλέον ε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ε, και άλλο να έχουμε το κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με τις αρμοδιότητες που μας έχουν δοθεί, να πείσουμε τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη, ότι μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική είναι το καλύτερο εργαλείο για να ε, νικήσουμε την κρίση που ταλαιπωρεί την Ευρώπη εδώ και χρόνια. Ε, συγγνώμη που μακρηγόρησα κυρία Πρόεδρε, αλλά πιστεύω ότι ένα τέτοιο θέμα αξίζει και ε, να επεκταθούμε λιγάκι στα πλαίσια του περιορισμένου χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας για τη συζήτηση αυτή. Θεωρώ όμως ότι η βιομηχανική πολιτική είναι ένα από τα θέματα ε, που έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Όλοι συμβάλλετε, ακόμα και με ε, σκληρές κριτικές και η συμβολή σας αυτή δείχνει πόση βούληση υπάρχει ε, για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής μας Κλείνοντας, ε, επιβεβαιώνω την τη δέσμευσή μου ότι θα κάνω ό,τι ε, περνάει από το χέρι μου για να ξαναγίνει η ε, ε, Ευρώπη, για να αποκτήσει μια μηχανική πολιτική, σίγουρα διαφορετική από τη δεκαετία του 50, αλλά πάντα στην πρωτοφορία όσον αφορά την ποιότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, λέει η Πρόεδρος. Ας περάσουμε τώρα στις παρεμβάσεις του ενός λεπτού. Ε, do la parola all'onorevole ε, Diaz de Mera. Diaz de Mera, παρακαλώ. La empresa Soriana Puertas Normas. Έχουμε μία επιχείρηση της Σόρια που έχει έδρα στην Ισπανία